Iniziamo. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Benvenuti. Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς επιστρέψατε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι ξεκουραστήκατε και είμαι επίσης βέβαιος ότι θα έχουμε ένα φθινόπωρο το οποίο θα είναι πολύ γεμάτο ε, με πολλή δουλειά και με πολλές υποχρεώσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Εάν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις από του σχεδίου μερσίας διατάξεως θεωρείται ε, εγκεκριμένο. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε διερμηνία σήμερα σε όλες τις γλώσσες εργασίες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα επίσης ε, για να κάνω κάτι που δεν κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή δεν είχαμε την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για την πολύ σημαντική συνάντηση αποστολή που είχαμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές από τις 14 μέχρι τις 17 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια αποστολή στην οποία εκτός από τον Πρόεδρο συμμετείχαν εννέα άλλοι συνάδελφοι. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της αντιπροσωπείας είχαμε συναντήσεις σε πάρα πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο. Συναντήσαμε τον Υπουργό Γεωργίας, Τόμ Βίλσακ, τον εκπρόσωπο εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Ρον Κίρκ καθώς επίσης την πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, Γεωργίας της ε, Γερουσίας, την κυρία Ντέμπι Στάμπενάου. Επίσης, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και συζήτηση στις Ηνωμένες, στα Ηνωμένα Έθνη με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Ρόμπερτ Ορ, καθώς επίσης και εκπροσώπους των μεγαλύτερων οργανισμών που ασχολούνται με την διατροφική ασφάλεια, όπως τον ΦΑΟ, το World Food Program κλπ. Γνωρίζετε φαντάζομαι ότι ε, ξεκινά και στις ΗΠΑ μια μεταρρύθμιση της Farm Bill του νομοσχεδίου λοιπόν ε, για την ε, γεωργία και βρήκαμε πολλές αντιστοιχίες με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Επομένως ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία προβλέπονται στην Farm Bill, κυρίως δε όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με την λειτουργία της αγοράς, με τα προγράμματα διατροφής όπως ας πούμε το SNAP, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα ε, συμπληρωματικής βοήθειας ε, στην ε, διατροφή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο μουτάτης μουτάντης ρωμιάζει με το δικό μας πρόγραμμα βοήθειας. Όμως πρέπει να πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες 70% όλου του προϋπολογισμού για την γεωργία απασχολείται από προγράμματα τέτοιου είδους και αφορά ακριβώς την βοήθεια βοήθεια πολιτών που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα επιβίωσης. Επίσης, είχαμε ε, συναντήσεις ε, και με την, ε, με την αντίστοιχη πλευρά των ΗΠΑ για τα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημεία τριβής μεταξύ των πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρέθη η λύση όσον αφορά τις ορμόνες στο βόλιο κρέας. Μιλήσαμε πάντως και για το βόλιο κρέας, αλλά μιλήσαμε και για άλλα ευρωπαϊκά δικά μας ε, συμφέροντα. Μιλήσαμε με τον Τόμ Βίλσακ αλλά και με τον Τόμ ε, Κίρκ, τον ε, εκπρόσωπο λοιπόν του εμπορίου, το ζήτημα το οποίο αφορά την επίλυση του προβλήματος των εξαγωγών κρέατος προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μετά τη σπονγκόδη κεφαλοπάθεια δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ελπίζουμε ότι αυτή η σημαντική αποστολή θα μπορέσει να ε, μας βοηθήσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Είχαμε επίσης ε, την ευκαιρία ε, να πάμε στην Barber's Vineyard που είναι στην περιοχή της Ουάσιγκτον μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ένα πολύ ενδιαφέρον χτήμα έτσι ώστε να δούμε ακριβώς πόσο δουλεύουν ε, οι νοπαραγωγοί στις ΗΠΑ. Τέλος, όπως σας είχα πει και αρχικά, ε, ολοκληρώθηκε η ε, επίσκεψη της με μια συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί συζητήθηκε ο ρόλος τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς επίσης και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση των ιδρυτικών προβλημάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτά επανειλημμένα ανεφέρθησαν και από την δική μας πλευρά, αλλά και από τα Ηνωμένα Έθνη. Βεβαίως, ενδεχομένως ενδεχομένως μετά από αυτήν ε, την αποστολή στις ΗΠΑ ενδεχομένως δεν αποκλείομαι ε, να έχουμε και ε, συναντήσεις πλέον στο δικό μας έδαφος με, από άτομα τα οποία συναντήσαμε στις ΗΠΑ. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3. Η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο για όλα τα τμήματα. η συγητής και συντάκτης μάλλον της γνωμοδότησης είναι ο Λουίς Καπούλος. Ε, Τζιμ, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, εγώ θα ήθελα όμως ε, να ε, αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια του ε, ε, καλοκαιριού. Φαίνεται ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού συστηματικά ε, είχαμε διάφορες αλλαγές. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πολλές διαρροές δηλαδή. Αυτές οι διαρροές δεν είναι δυνατόν να είναι όλες κατά λάθος γιατί ε, είχαμε πολλές διαρροές όσον αφορά συγκεκριμένα σημεία των ε, νομικών κειμένων ε, που θα κοινοποιηθούν και θα γνωστοποιηθούν τον Οκτώβριο. Εν πάση περιπτώσει μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροδιαρροές δεξιά-αριστερά, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς ολόκληρο το έγγραφο στο, στα χέρια του. Επομένως θέλω μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πάντα προσπαθούν να παρακάμπτουν την Επιτροπή μας, γιατί πάντα κοινοποιούνται τα πάντα στην κοινή γνώμη, δημοσιοποιούνται όλα, πριν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Ε, κοιτάξτε, η δικιά μας ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, αυτά τα θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας είναι από τα πιο σημαντικά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από τη δικιά μας δουλειά εξαρτώνται εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Επομένως, εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει αν η Κομισιόν κάνει καλά τη δουλειά, τους, τη δουλειά αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Και επομένως αυτές οι διαρροές είναι απαράδεκτες από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, σας ερωτώ ευθέως, γιατί πάντα ε, κοινοποιείτε σε όλο τον κόσμο διάφορα πράγματα σχετικά με τη γεωργική πολιτική πριν και χωρίς να μιλήσετε στη δική μας Επιτροπή. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει μια γενική διεύθυνση η οποία προσπαθεί να τα κάνει πλακάκια κατά κάποιο τρόπο με τα μέσα ενημέρωση τα οποία ασχολούνται με τη γεωργία. Ε, δεν ξέρω εάν ε, υπάρχει μια γενική διεύθυνση που προσπαθεί να υποσκελίσει μια άλλη γενική διεύθυνση και στο τέλο δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Όλη αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει εμεί, σαν ε, Επιτροπή του Κοινοβουλίου να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα για το θέμα. Αυτό ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε ε, την άποψή σου και μάλιστα και στην ε, διάρκεια ε, ξέρετε, των διοργανικών συζητήσεων. Καμιά φορά ε, μπορεί να υπάρξουν τέτοιου είδους ε, ατυχήματα. Εν πάση περιπτώσει όμως συμφωνούμε, συμφωνούμε με όλα αυτά και το λαμβάνουμε υπόψη μας. Προχωράμε πάντως στο σημείο 3, λέγαμε ότι είναι η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Μετά τη συζήτηση θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες οι οποίες ε, έχουν ε, υποβληθεί στο σχέδιο προπολογισμού 2012 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο. Η ψηφοφορία επί του κειμένου της ε, γνωμοδότησης θα γίνει αργότερα το Σεπτέμβριο. Ε, Πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες ε, τροπολογίες έχουν λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τροπολογίες επίσης οι οποίες ασχολούνται ε, με την ε, πρώτη φάση ή τη δεύτερη, ή τη δεύτερη φάση. Υπάρχουν άλλες οι οποίες ασχολούνται με τις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Σε πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ όλα αυτά. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος να σας τα πει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιστροφή σε όλους τους συναδέλφους, καλή δουλειά. Ελπίζω να ξεκουράστηκαν στις διακοπές τους, γιατί χρειαζόμαστε δύναμη για τις μελλοντικές μας εργασίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδους ηγητές, καθώς και όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν προτάσεις και τροπολογίες και ευχαριστώ και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαθεσιμότητά τους. Μας βοήθησαν για να διαλευκάνουμε διάφορες αμφιβολίες που είχαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η πρόταση του Συμβουλίου ε, συνιστά μια ουσιαστικότατη μείωση σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με τα ε, ταμεία των παραγωγών για τα απορροκυπευτικά, για τη διανομή στα σχολεία φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόκληση των απόψεων ανάμεσα στον εισηγητή μου δηλαδή και την πρόταση και τις του Συμβουλίου. Ε, όπου δεν λαμβάνεται υπόψη οι αρχικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, το Συμβούλιο... Ε, λοιπόν, κάνει μια πρόταση που δεν είναι ρεαλιστική όπως της Επιτροπής. Ε, και διαφέρει αυτό πολύ σε σχέση με το μέσο όρο των δαπανών των περασμένων ετών. Ε, πολλές ε, από τις τροπολογίες, όπως είπε και ο Πρόεδρος μας, σχετίζονται με τον αρχικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εξάλλου προτείνω και εγώ μέσα στην έκθεσή μου και προτείνω λοιπόν να συμπεριλάβουμε διάφορες προτάσεις που συνεπάγονται αυξημένες δαπάνες, όπως ε, η αποζημίωση παραδείγματος χάρη των γεωργών ε, που ε, επλήγησαν από το βακτηρίδιο ή κόλλη ε, επίσης θέλω να αναφερθώ στα προγράμματα πιλότους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά τα προγράμματα και ταυτόχρονα ε, προτείνω απόρριψη αυτών που σχετίζονται με θέματα που βραχυπρόθεσμα θα συζητηθούν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε η πρόταση που καλούμε τώρα να εγκρίνουμε νομίζω θα βελτιωθεί με τις τροπολογίες ε, που θα προσθέσω στο κείμενο και θα ε, συνιστά μια καλή βάση για τις μελλοντικές εργασίες μας για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ελπίζω η Επιτροπή Προϋπολογισμών να δεχτεί την συνεισφορά της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Λουίς. Ε, εάν δεν ζητάει κανείς το λόγο, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι φαντάζομαι τις κάρτες σας. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, προτείνω να ψηφίσουμε on block ομού όλες ε, τις ε, ε, τροπολογίες οι οποίες αφορούν την κατάσταση πριν από την τροποποίηση του Συμβουλίου. Πρόκειται για έξι τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiaro chiusa la votazione. Πέρας. Quindi in blocco abbiamo... Ωραία. Ε, σαφώς εγκρίνονται. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 5226. Πιλωτικό πρόγραμμα Νέα Γραμμή, άρχεται η ψηφοφορία 5226. Πέρας. Εγκρίνεται νομίζω, ναι, εγκρίνεται. 52-28. Παρακαλώ. Λουίς. Ζητώ συγγνώμη αλλά ε, δοθεί τη δυσκολία ε, συγκέντρωση μετά τι διακοπέ. Διαπιστώνω ότι δεν έχω την κάρτα μου μας, την ηλεκτρονική κάρτα και δεν είμαι και ο μόνο νομίζω. Παρακαλώ, προσθέστε τι ψήφου μα, ε, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίω θα λάβουμε υπόψη μα τι ψήφου σα, αλίμονο. 52-28 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε. 52, στην 52-72, τροπολογία 52-72, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 52-72 απορρίπτεται. Επόμενη τροπολογία 52-65. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 52-65. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. 52-79. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 52-79. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στο 52, στην 52-41 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Νομίζω πως εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. 52-80 Άρχεται η ψηφοφορία επί της 5280. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 5273. 5273. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5268, 5268, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5275. 5275 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 52-45, 52-45, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία Τροπολογία 52-69, 52-69, Άρχεται η ψηφοφορία 52 52-69. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Πέρας, εγκρίνεται. Και τώρα τι θα ψηφίσουμε. «5281». 5281. 5281. 81 αρχεται η ψηφοφορία επί της 52-81. Πέρας. Εγκρίνεται. 5271, τροπολογία επί της τροπολογίας 5271, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 5223, 5223, πέρας της ψηφοφορίας, Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία 5266. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 5266 πέρας. Της ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 5266. 52-51 πρέπει να τη σελίδα. Είναι η τροπολογία 52-51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα η τροπολογία 52-52. Άρχεται η ψηφοφορία 52-52. Πέρας και εγκρίνεται. Πενήντα εξήντα 52-67 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κάτι, κάποιος δεν ψήφισε. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 52-32, 52-32. Έχετε κάτι να πείτε? Παρακαλώ κύριε Λάγκη. Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Πρώτα για τις γενικές παρατηρήσεις λοιπόν όσον αφορά την σημασία αυτής της έρευνας και μετά ψήφο ε, που θα αφορά την διεύρυνση του ε, πεδίου που θεωρούμε σαν ΕΛΚ ότι ε, εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί ήδη ε, ε, κοπιάζουμε για να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα. Πολλό δε μάλλον... Ωραία, δει και δίκιο κυρία Ντελάνς, 52-32 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, πέρα της ψηφοφορια δεν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε 52-32 δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 52-32. Για να δούμε. Απορρίπτεται το δεύτερο. Τροπολογία 5234. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 5234. Πέρας. Απορρίπτεται. 5227. Άρχεται η ψηφοφορία. 5227. Πέρας της ψηφοφορίας επί της 5227. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Κατά λάθος ο πρόεδρος είπε απορρίπτεται. Εγκρίνεται. 52-24. 52-24. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και πού θα πάμε τώρα σε ίδια 52 52-74. Ψηφίζουμε επί της 52-74. Πέρας απορρίπτεται. 5270. 5270. 5270 άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5270. Πέρας. Απορρίπτεται. 5231 άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5231. 5231. Απορρίπτεται και αυτή η τροπολογία μάλλον λέει ο Πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας πάντως. Ορίστε. Απερίφθη. 52-30. 52-30. Άρχεται η ψηφοφορία. 52-30. Πέρας της ε, ψηφοφοριας απολυπτεται απορρίπτεται. 52-25. 52-25 άρχεται η ψηφοφορία. 52-25. Πέρας της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. 52-29. Ψηφίζουμε επί της 52-29. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 52-57. 52-57 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. «52-76», «52-76», εγκρίνεται νομίζω, λέει ο Προεδρο. πέρας τη ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται, ορίστε, Σα το είπα. Εγκρίνεται το 5276. 5278. 5278 άρχεται η ψηφοφορία. 5278 πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. τώρα θα ψηφίσουμε. 52-13. 52-13. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. 52-13. Άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας. Είμαι σίγουρος ότι έχει εγκριθεί. 52-77. Άρχεται η ψηφοφορία. όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι είναι έκτακτο αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορεί ορισμένοι να υπομοιδιάσουν, δεν ξέρω, αλλά θα σας παρακαλούσα το εξής. Με την άδειά σα, βέβαια, μια προφορική τροπολογία να ψηφίσουμε. Βεβαίω, 05, 08, 06 είναι το κονδύλι. Ξέρω ότι είναι δεχομένως πιλωτικό πρόγραμμα, αλλά σκοπός είναι να ενισχυθεί ένα δίκτυο για την προστασία της οικογενειακής γεωργίας στην Ευρώπη. Ε, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία αλλά και στην Ελβετία πολλές οργανώσεις εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και θα θέλαμε η Πολωνία και η Πορτογαλία να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο έτσι σε ευρικό στάδιο θέλετε αλλά και ε, αργότερα άλλα κράτη γιατί παντού έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ε, φτωχεύουν οι γεωργοί, δεν θα σας δώσω ε, στοιχεία, αλλά για τις τέσσερις χώρες, Γαλλία, Γερμανία, επαναλαμβάνω, Γερμανία ε, και Ελβετία, είναι τέσσερα ε, τα σωματεία με 98 εργαζομένους που εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Ακούμε τα προβλήματα στη Γεωργία, αυξάνονται οι αυτοκτονίες, έτσι, και όχι μόνο. Και γενικά μεγάλη απόγνωση, πίκρα στην Ήπεθρο. Και πριν από τις διακοπές Είχαμε συναντηθεί με διάφορους ενδιαφερομένους και μετά μας είπαν «Α, τώρα όμω θα φύγουμε για διακοπές». Γι' αυτό προτείνω την προφορική τροπολογία και πρόκειται για 348.000 πέρα από το σχέδιο προϋπολογισμού να προσθεθούν αυτά στο 050806 μπορεί να είναι πιλωτικό πρόγραμμα και θα δούμε στη συνέχεια. Αν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία, απευθύνομαι σε όλες τις πολιτικές ομάδες, διότι οι σκιώδες ηγητές έχουν ειδικό βάρος. Και την κυρία Ντελάγκε και από πίσω της τον κύριο Σιλβέστρης κοιτάω. Ε, αυτός φαντάζομαι θα με ιδιάσει όπως έλεγα προηγουμένως με το έτοιμά μου. Αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά γνωστή. Μπορεί κάτι να φαίνεται θεμητό. Ε, ξέρω ότι ε, κάπως αποκλίνει από τις διαδικασίες. Δεν θέλω να γίνει κανόνας, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερη η περιστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπέλα. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση προφορικής τροπολογίας. Ξέρετε ποιοι είναι οι κανονισμοί, αν συμφωνούμε όλοι. Ναι, θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ντελάγκη. Απλώς έλεγα ότι για να εγκριθεί μια προφορική τροπολογία θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να αντιτίθεται στην ιδέα αυτή. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ντελάνγκε, παρακαλώ, και μετά στον Σιλβέστρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω τα προγράμματα αυτά πάρα πολύ καλά και βεβαίως γνωρίζουμε ότι διανύει πολύ δυσχερή περίοδο η Γεωργία. Έχουμε επίσης και μια τηλεφωνική γραμμή την οποία μπορούν, στην οποία μπορούν να ζητήσουν βοήθεια οι Γεωργοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω κύριε Ταραμπέλα την σημασία των προγραμμάτων αυτών. Από την άλλη πλευρά όμως είμαστε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επομένως βεβαίως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 δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι εύκολα το οποίο αναφέρεται σε πέντε χώρες και όχι σε 27. Ε, κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε βεβαίως ε, συμβιβαστικές λύσεις ε, χωρίς πολύ πολύ κουβέντα. Επομένως, ναι, συμφωνώ με την ιδέα, αλλά θα ήθελα να τη διατυπώσετε με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στους 27 και όχι στους 5. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είχε δει στο λόγο? Σιλβέστρης? Όχι. Όχι. θα ξαναδώσω το λόγο στον ε, Μάρκ Ταραμπέλα για να απαντήσει σε αυτή την παρατήρηση. Πολύ σύντομα, ναι, βεβαίω συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Ντελάγκε και φυσικά προσυπογράφω όλα αυτά που είπε. Ε, είναι γεγονό ότι σε ορισμένε από τι χώρε αυτέ τι οποίε ανέφερα ε, υφίστανται ήδη κάποιε υπηρεσίε βοήθεια. Γνωρίζομαι βεβαίω ότι τα προβλήματα ε, του γεωργικού κόσμου αφορούν όλε τι χώρε. Εδώ αυτό που προτείνω εγώ είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εμβριακή Α το πούμε κατάσταση που ελπίζουμε ότι θα μεγαλώσει και θα αφορά πλέον όλες τις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, είτε ε, βασίζομαι στην ιδέα αυτή και λέω ότι εάν κάποιες χώρες έχουν ήδη κάποιες τέτοιες υπηρεσίες τότε να τις διευρύνουν, ενώ άλλες να πάρουν ιδέες έτσι ώστε να δημιουργήσουν τέτοιες υπηρεσίες αρρωγής των γεωργών. Κυρία Ντελάγκε. Οι άντρες οι οποίοι μιλούν γαλλικά είναι πάντοτε εξαιρετικά ελκυστικοί. Παρόλα αυτά εγώ θα αντισταθώ. Ε, Κοιτάξτε, ε, είπαμε, εάν προσθέσετε και άλλες χώρες ε, ή αν βγάλετε τις, ε, την συγκεκριμένη αναφορά στις πέντε ε, χώρες, τότε παρά την μεγάλη γοητεία που είχε αυτή η γαλλική σας εισαγωγή εγώ θα αντισταθώ. Πιστεύω ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές ε, τις ιδέες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τότε πραγματικά θα σας στηρίξω. Ε, ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ με την πρόταση της κυρίας Ντελάγκ. δηλαδή να μην ε, γίνει αναφορά ονομαστική στις χώρες οι οποίες έχουν ήδη είτε ένα πιλωτικό τέτοιο πρόγραμμα, είτε ε, έτσι μια ιδέα τέτοιου προγράμματος. Να αφαιρεθούν λοιπόν ε, αυτά τα, αυτές οι χώρες ε, και αν συμφωνεί και ο Μάρκ τότε νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την προφορική τροπολογία. Διαφορετικά θα έχουμε δυσκολία. Θα ήταν ένα πρώτο βήμα συνάδελφοι είμαστε, κανείς δεν αντιτάχθηκε σε αυτή την αρχή, το θέμα είναι να περάσει το μήνυμα, αλλά πρέπει να δούμε και τι μας δείχνει η εμπειρία, δεν υπάρχουν ακόμα όλα αυτά τα δίκτυα και οι επαφές, οπότε ναι, εντάξει, γοητευτικά είναι τα γαλλικά, αλλά Netherlands OK. Και τα Ολλανδικά, μπορώ να σα τα πω και Ολλανδικά θέλετε. Δεν είναι η μητρική μου, αλλά την κατέχω. Εν πάση περιπτώσει, με τα Ολλανδικούλια μου μπορώ να σα τα πω για να είμαι ακριβή. Γι' αυτό συνεχίζω όμω στα γαλλικά, γιατί θέλω να είμαι ε, ακριβής. Στα Ολλανδικά δεν μπορώ να το πω τόσο. Ε, ε, μιλάμε για ένα σχέδιο. Όποιο θέλει μπορεί να μπει σε αυτό το σχέδιο, το πιλωτικό πρόγραμμα. Αν είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μπει. Και δεν θα απορρίψουμε του Ελβετού, ε, γιατί έχουν και εκείνη πείρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι στην αυλή μα. Αυτά. Νομίζω ότι είναι καλή συμβαστική πρόταση. Αυτή είναι η ιδέα, εν περιπτώσει. Άψογα με την ε, τροπολογία λοιπόν έτσι όπως την αποσαφήνισε η κυρία Ντελάνγκε, χωρίς να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες χώρες ψηφίζουμε αυτή την προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με τη διόρθωση λοιπόν της κυρίας Ντελάνγκε. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Andiamo aperto il voto al 52-77. 52-77 άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione, direi... Πέρας, νομίζω ότι θα έχει εγκριθεί. Καλά μάντεψα. 52-22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, πέρας της ψηφοφορίας από της ε, τροπολογίας 52-22. Εγκρίνεται. 52-12, άρχεται η ψηφοφορία επί της 52-12, πέρας, πέρας, νομίζω πως θα εγκριθεί και αυτή, εγκρίθηκε, τέλος, 52-00, 52-00 άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ, πέρας, εγκρίνεται. Τέλος. Α, όχι, δεν, δεν υπάρχει τέλος, δεν έχουμε τελική ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Και επομένως ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφιση των τροπολογιών αυτών. Σας υπενθυμίζω όμως ότι όσον αφορά τι τροπολογίες επί του κειμένου, η προθεσμία υποβολής είναι η 5η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ όλους. Περνούμε τώρα στο σημείο 4 της ημερησίας διατάξεως. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού 1698 κάθετο 2005 του Συμβουλίου όσον αφορά κάποιε διατάξει που σχετίζονται με τη δημοσιονομική διαχείριση για κάποια κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίε ή απειλούνται ε, με σοβαρέ δυσκολίε σε σχέση με την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, λαμβάνοντα υπόψη τις ε, σοβαρές ε, χρηματοοικονομικές δυσχέρειες τις οποίε αντιμετωπίζουν κάποιε χώρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία πρόταση ε, που αφορά την ε, ε, μείωση της συνεισφοράς για κάποια προγράμματα γεωργικά 85 ή 95 στο 85 στο 95% για το 2011 και για το 2012. Όμως τα επιχειρησιακά προγράμματα του 2007-2013 του ΦΕΟΓΚΑ δεν θα επηρεαστούν. Ε, σήμερα το απόγευμα με τους συντονιστές θα ορίσουμε ε, και αυτόν που θα ασχοληθεί ε, με το θέμα. Τώρα, στρέφουμε προς την Επιτροπή, αλλά είναι εδώ η Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Αναμέναμε την δόκτωρα Ντόρμαν Μαρίνο, αλλά δεν τη βλέπω να έχει έρθει. Α. Ναι, νομίζω ότι έχουν λίγο αργοπορήσει οι συναδελφοί μου, αλλά πάντως θα καλύψω με το κενό της απουσίας τους, γιατί έρχονται όπου να είναι. Νομίζω ότι η ίδια η πρόταση είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτα απ' όλα, Το πνεύμα της ε, πρότασης νομίζω είναι ε, σαφές. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. Και δεν μπορώ να πω ότι έχουμε άλλες παρατηρήσεις να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ίσως εμείς προχωρήσαμε με πολύ ταχυριθμό και γι' αυτό δεν έφτασε η εκπρόσωπος. Εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως ε, η παρουσίαση θα ήταν πάρα πολύ συνθετική. Ξέρετε ποια είναι τα προγράμματα ανάπτυξης της επέθρου, ξέρετε ποιες είναι οι δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν ε, οι χώρες αυτές και επομένως έγινε η πρόταση να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και άλλες ενδεχομένως ε, χώρες. Ε, ο, η Μάριαν έχει ζητήσει το λόγο όμω, Μάριαν Μαγκίνε, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα παρουσιάσει κάποια παραδείγματα στην πράξη. Τι γίνεται, όπω είπε και ο Τζιν Νίκολσον, ε, για τη διαρροή των εγγράφων που δημιουργούν αυτή τη σύγχυση και τι ανησυχίε, Έτσι και εδώ ε, έχει δημιουργήσει έντονε συζητήσει ε, αυτή η πρόταση γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιπρόσθετα κονδύλια. Εγώ από ό,τι έμαθα όμω, δεν υπάρχουν αυτά ε, ίσως είναι θέμα ε, ε, ε, εκταμίευσης των κονδυλίων, πρόορης εκταμίευσης των κονδυλίων. Οπότε θέλω να μάθω, οι χώρες που έχουν δυσκολίες πώς θα επηρεαστούν. δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουν κάποια μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπέρ άλλων. δεν, δεν έχω καταλάβει καθόλου περί τίνος πρόκειται. Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις αυτής της νέας της πρότασης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο σχέδιος εισηγητής... Α, όχι, η, ο κύριος Παπαστάμκος. Ο κύριος Παπαστάμκος ζητάει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ε, συμφωνώ με την ε, κυρία Μαγκίνες ότι ε, πρέπει να ξέρουμε το διαγραφόμενο πλαίσιο αυτής της ελάφρυσης χωρών οι οποίε αντιμετωπίζουν ε, την, κρίση, τις συνέπειες της κρίσης και θα μπορούσε ίσως η, Επιτροπή να φωτίσει ακόμη περισσότερο και σε αυτό το στάδιο ε, με τις ε, δικές της ιδέες, σκέψεις ε, και προτάσεις για να γνωρίζουμε προς τα πού βαδίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δανέλης επίσης έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα χαιρετίζω την ε, πρόταση της Επιτροπής γιατί δείχνει ότι με ευαισθησία αντιλαμβάνεται τις δύσκολες ε, συγκυρίες που κάποιες χώρες και η λαοί της και ιδιαίτερα η αγροτική τάξη αντιμετωπίζει σε αυτή την περίοδο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω την Επιτροπή αν συμφωνεί ότι αφού θα έχουμε μείωση του συνολικού προϋπολογισμού που θα διατεθεί αν θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένη να υπάρξει μία, ε, μία διευκόλυνση και στα ζητήματα της τροποποίησης των σχεδιασμών που θα ακολουθήσουν ε, και όσον αφορά τους χρόνους και όσον αφορά τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σπύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί της αρχής η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακούγεται λογική και σωστή. Έχω συμπληρωματικέ ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε στα χέρια μας το έγγραφο συγκεκριμένα. Τρεις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ποιος ορίζει τη δυσχερή θέση, πώς ορίζεται αυτό, ε, ε υπολογίζεται, ποια είναι αυτή η περίπτωση, πότε θα εμφανιστεί με κάποια στοιχεία αριθμητικά είναι πολιτική απόφαση. Πώς ορίζεται αυτή η δυσχέρεια και για ποιον ισχύει αυτό συγκεκριμένα. Μετά ισχύει για όλα τα προγράμματα ή μόνο για ορισμένα η δεύτερη ερώτηση. Και ερώτηση τρίτη. Για αυτή την ε, περίπτωση. Πώς να το πω. Θα αυξηθεί η ευρωπαϊκή συμμετοχή Και αυτό δεν σημαίνει στη συνέχεια θα είναι και πιο ε, πυκνή η έλεγχη, θα είναι περισσότερη έλεγχη για την εφαρμογή και αν πιάνουν τόπο αυτά τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ. Ε, η κυρία Ρέιμετς. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ και εγώ με τις ερωτήσεις του κυρίου Γιάρ, αλλά έχω και μια άλλη ερώτηση για να καταλάβω. Αν η ανάληψη υποχρεώσεων δεν αυξηθεί, δεν είναι περισσότερα τα χρήματα προπολογισμού, αλλά παρόλα αυτά δίνουμε περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθηματικά δεν μου βγαίνει, δεν το καταλαβαίνω. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Ε, θα κάνουμε οικονομίες από αλλού, αν ναι από πού και πού υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνουμε οικονομίες. Τι, μήπως είχαμε μέχρι τώρα τίποτα λεφτά που δεν τα απορροφούσαμε και θα τα δώσουμε εκεί, δεν το καταλαβαίνω. Με ξεπερνάει. Πού θα, όπου βρίσκουμε ξαφνικά λεφτά. Εγώ επειδή είμαι και επιχειρηματίας δεν καταλαβαίνω πού τα βρήκαμε ξαφνικά. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό έχει έρθει ο δόκτωρ Άλντο Λόγκο να μας τα εξηγήσει και να μας τα πει όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων και των γνώσεών μου να υποκαταστήσω την ε, ε, δόκτωρα Μαρίνο η οποία θα φτάσει σε λίγο. Η πρόταση αφορά κυρίως την δυνατότητα η οποία δίνεται σε κάποια κράτη-μέλη, κυρίως δεν σε πέντε χώρες-μέλη, να αυξήσουν το ποσοστό ε, ε, συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου που χρηματοδοτούνται από το ΦΕΟΓΑ. Αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το μέγιστο του 95% στις ζώνες σύγκλησης στις ε, νήσους του Αιγαίου επίσης, επίσης και ε, μπορεί να φτάσει μέχρι το 85% στις υπόλοιπες περιοχές. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι ο συνολικός όγκος της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν αλλάζει. Οι πόροι είναι αυτοί που είναι, είναι αυτοί που εξ αρχής έχουν δοθεί ε, στις, στα προγράμματα αυτά. Όμως μειώνεται το ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης. Αυτή είναι η δυνατότητα η οποία δίνεται στις χώρες μέλη έτσι ώστε ε, να ανακουφιστούν κατά κάποιο τρόπο τα δημόσια οικονομικά των χωρών αλλά ταυτοχρόνως να στηριχτούν, να βοηθηθούν οι εν λόγω περιοχές γιατί τα χρήματα στο σύνολό τους που θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση των ελόγων προγραμμάτων θα είναι ε, λιγότερα εξακολουθώ και το ξαναλέω ότι ο όγκος των χρημάτων από τη μία και την άλλη πλευρά ε, δεν ε, αλλάζει, δηλαδή ε, μάλλον τροποποιείται μονάχα το κομμάτι της εθνικής χρηματοδότησης. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά σημεία τα οποία ακριβώς αποτελούν την πρόταση. Θα ήθελα επίσης να αποσαφηνίσω και κάποια άλλα σημεία τα οποία εφήγησαν εδώ και για τα οποία νομίζω ότι ε, η δόκτωρ ε, Μαρίνο θα μας δώσει τις ε, απαντήσεις σε λεπτομέρεια γιατί την είδα ότι φτάνει. Την είδα λίγο στην πόρτα. Πάντως υπάρχει ένα σημείο το οποίο αφορά το εξής, δηλαδή ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο γενικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού. Αυτό το γενικό αντίκτυπο δεν μπορούμε να τον ποσοστοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένους αριθμούς, όμως μπορούμε να κάνουμε κάποιες γενικές εκτιμήσεις που θα αφορούν την συνολική θετική επίπτωση αυτού του μέτρου. Θα δώσω τώρα το λόγο αμέσως στην συνάδελφό μου η οποία είναι σε θέση να αποσαφηνίσει περαιτέρω λεπτομέρειες της εν λόγω πρότασης. Ευχαριστώ πολύ δόκτωρα Λόγκο, χαιρετίζω την ε, δόκτωρα Μαρίνο αλλά θα δώσω ξανά τον ε, λόγο στην κυρία Μαγκίνες και σε έναν άλλο συνάδελφο που ζήτησαν τον λόγο. Μάριον, ζήτησες ξανά τον λόγο. Ευχαριστώ. Μπορεί να ε, αυτή οι διακοπές και να είμαι αργή ακόμη, αλλά πρέπει να είμαστε σαφέστεροι κατά τη γνώμη μου. Τι ισχύει. Ε, θα δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη-μέλη σε κάποια προγράμματα ούτως ώστε το συνολικό ποσό κατανέμεται σε λιγότερα προγράμματα διότι αν παραμείνει ίδια, ίδιο το ποσό αλλά αυξηθεί το ποσοστό της χρηματοδότησης θέλω ε, να το καταλάβω. Πείτε με χαζή, πείτε με αργή, πείτε με ό,τι θέλετε. Θέλω να καταλάβω. Ε, Μπορεί να υπάρχει μια απλούστατη εξήγηση, απλώ ακόμη δεν την άκουσα. Θέλω να μάθω στην πράξη τι ισχύει. Τα κράτη-μέλη που πλήττονται από αυτό ρωτούν το εξή. Θα δοθεί προτεραιότητα σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα ή για κάποιε χώρε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ε, και προτείνεται αυτό το νέο σύστημα. Ε, θέλω να αιτιολογήσετε αυτή στην πρόταση. Ευχαριστούμε, κυρία Ρέμε. Ευχαριστώ πολύ. Το ίδιο θα πω κι εγώ. Ότι είναι ίδιο το ποσό λέτε, αλλά η συγχρηματοδότηση, η συνυπευθυνότητα του κράτου μέλους μειώνεται. Άρα είναι λογικό ότι είναι λιγότερα τα προγράμματα. Η πρώτη ερώτηση είναι και τι βοηθάμε, έτσι. Και η δεύτερη ερώτηση, δεν θα είχε περισσότερο νόημα να βοηθήσουμε λιγότερα προγράμματα παρά καθόλου τίποτα. Αυτή η ιδέα μας έχει προβληματίσει. Αυτό κρύβεται από πίσω. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει με ποιο συλλογισμό έχει καταλήξει σε αυτή την πρόταση. Λουίς. Λουίς Κάπουλα Σαντός, Ο Λουίς Κάπουλα Σάντος έχει ζητήσει το λόγο και μετά θα ακούσουμε την ε, κυρία Μαρίνο. Ε, πρόεδρε, ε, εκπλήσωμαι από το ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι τόσο δυσνόητη για κάποιους συναδέλφους. Θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση. Φανταστείτε, ένα κράτος όπου υπάρχουν δημοσιονομικές δυσκολίες και όπου χρειάζονται περικοπές, δραστικές περικοπές στην παιδεία, στην υγεία, ε, στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι προφανές λοιπόν ότι όταν χρειάζονται τέτοιες ομές περικοπές στον προϋπολογισμό, η βασική τομή είναι εκείνοι όπου δεν μπορούν να γίνουν περικοπές. Η γεωργία λοιπόν προκύπτει ως μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά αν δεν υπάρχει ε, εθνική συγχρηματοδότηση, τα προγράμματα ανάπτυξης επέθρου δεν μπορούν ε, να ε, τροποποιηθούν. Αυτή η απόφαση τι στόχο έχει να επιτρέψει μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να λιγοστεύσει το ποσοστό συγχρηματοδότηση στο εθνικό και να συνεχιστούν τα προγράμματα. Ούτε Κατά ένα σεντ δεν ε, ε, ε, αυξάνονται τα κονδύλια. Τα προγράμματα ε, ανάπτυξης υπαίθρου πρέπει να εκτελεστούν στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι και τίποτα παραπάνω και ελπίζω ε, να μην αντιμετωπίσουν και άλλα κράτη-μέλη αντίστοιχη κατάσταση και να χρειαστεί να κινητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αλληλεγγύης. Αν προκύψει κάτι τέτοιο θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός. Αλλά ε, περί αυτού πρόκειται. Για ένα κράτος μέλος θέλουμε να, συνεχιστούν, να συνεχιστεί η εκμε εκταμείευση κονδυλίων μειώνοντα το ποσοστό, το εθνικό ποσοστό συγχρηματοδότηση. Αυτό και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον Λύ και τώρα θα ακούσουμε τον διευθυντή, τη διευθύντρια Μαρίνο. Thank you very much, Chairman, and please excuse... Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρησή μου. Νόμιζα ότι θα κρατούσε περισσότερο η προηγούμενη συζήτηση. Ε, λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στην ουσία και θα απαντήσω σε αυτές τις τρεις ε, ερωτήσεις της κυρίας Μαγκίνης, ε, της κυρίας Ρέμες και του κυρίου Σάντος. Δεν θα σημειωθεί καμία απολύτως αύξηση στον προϋπολογισμό. Αυτό που θα συμβεί είναι μείωση του εθνικού ποσοστού συγχρηματοδότησης. Αυτό προφανώς σημαίνει πως θα είναι λιγότερα τα προγράμματα, ναι, αλλά ταυτόχρονα για αυτά τα κράτη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσουν τα προγράμματα, λοιπόν για αυτά τα κράτη το νέο σύστημα σημαίνει θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και δεν θα χάσουν ε, χρήματα ε, από, μετά το πέρας της περίοδου νη συν 2 για τις πληρωμές και έτσι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της χώρας. Ε, θα ήθελα να πω και άλλα δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Πρώτον, υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να μειώσουν το εθνικό ποσοστό συγχρηματοδότηση. Δεν συνιστά αυτό η υποχρέωση. Είναι μια εναλλακτική λύση. Θα αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη κατά πόσο θα χρειαστούν, αν θα χρειαστούν αυτήν τη νέα εναλλακτική λύση. Και δεύτερον, υποθέτουμε ότι τα προγράμματα που θα πληγούν θα είχαν χρηματοδοτηθεί στην περίοδο 2014 έως 2015. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο ελπίζουμε ότι τα νέα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου ήδη θα τρέχουν. Οπότε, ε, εάν εξελιχθεί αίσια η διαδικασία, αυτά που θα χάσουν από πλευρά σε προγραμμάτων θα αναπληρωθούν ε, κατά πάσα πιθανότητα ε, στο νέο, στα νέα προγράμματα ε, ανάπτυξης της Υπέθρου. Και ξαναλέω, αυτή είναι μια δυνατότητα που έχει η Ελλάδα, ε, η Πορτογαλία, η Λετωνία, η Ρουμανία και η Ιρλανδία. Πρόεδρε, θέλετε να κάνω μια πληρέστερη παρουσίαση, θέλετε να απαντήσω ρωτής πείτε μου ακριβώς τι θέλετε να κάνω. Ελπίζω τώρα τα πράγματα να είναι σαφή στο νου όλων. Δεν μιλάμε για αύξηση του προϋπολογισμού. Ε, ό,τι έχει προβλεφθεί, έχει προβλεφθεί. Βεβαίως ε, θα υπάρξει επομένως κάποια μείωση των προγραμμάτων ε, και επομένως με τα ίδια χρήματα θα χρηματοδοτηθούν κάποια λιγότερα προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες αυτές να συνεχίσουν με τα προγράμματα αυτά με λιγότερη χρηματοδότηση χρηματοδότηση από τη δική τους πλευρά. Ε... Ο ζητώ συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε. Ποιο ορίζει την έκτακτη κατάσταση, θα πρέπει κάποιο να υποβάλει ένα αίτημα, είναι αυτόματο, είναι ανοιχτή η διαδικασία, μπορούν να προσθεθούν χωρίς να αφαιρεθούν, να αποχωρούν. Ποιο το ορίζει αυτό, πότε μπορεί μια χώρα να κάνει χρήση αυτή τη ρύθμιση. Δόκτωρ ε, Μαρίνο, έχει, είχε τεθεί ένα ερώτημα από τον ε, κύριο Γιάρ πριν φτάσετε εσείς. Ποιος ε, λοιπόν καθορίζει τον κατάλογο των χωρών, ποια τήρια βάση των οποίων επιλέγονται οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί στον κατάλογο αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες από αυτών των σημείων. Δεν μπορεί να επεκταθεί ο κατάλογος στο μέτρο που προβλέπεται αυτή η ρύθμιση μόνο για τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν την ε, υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Δηλαδή μιλούμε για την ε, χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση, τη FSF και αυτό σχετίζεται με το ισοζύγιο πληρωμών και πρόκειται για μεσοπρόθεσμη χρηματοπιστωτική στήριξη ε, προς αυτά τα κράτη-μέλη Προηγουμένω ίσχυε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης. Τέλος πάντων αυτά τα κράτη-μέλη που είναι αποδέκτες της βοήθειας από τον ε, μηχανισμό, από το σύστημα μάλλον χρηματοπιστωτικής ε, σταθεροποίησης είναι επιλέξιμα αν θέλετε για αυτή, την, ε, για αυτή τη νέα ρύθμιση. Α, τα ίδια τα κράτη-μέλη, το τονίζω, θα αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εναλλακτική λύση. Αν ναι, θα χρειαστεί να υποβάλουμε πρόταση τροποποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης τη υπαίθρου και φυσικά ταυτόχρονα θα μεριμνήσουμε ώστε η πρόταση αυτή να μην υπονομεύσει τη συνολική στρατηγική και τους στόχους αυτής. Η πρόταση αυτή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να διαταράξει την ισορροπία στην οποία καταλήξαμε στο παρόν σύστημα ε, προγραμμάτων ανάπτυξης ε, της υπαίθρου. Προσβλέπουμε στη συζήτηση, στο διάλογο με αυτές τις χώρες, ε, μόλις το θέλησουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά ο κύριος ε, Χάσουρτ έχει ζητήσει το λόγο εν μεταξύ. Πρόεδρε, δύο ζητήματα που αφορούν και τα δύο τη διαχείριση των προγραμμάτων. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας σχολιάσει τι θα κάνει για ε, τη μελέτη αντικτύπου αυτών των μέτρων. Έχει γίνει, αν όχι προτείνουν να γίνει. Δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι πολλές από τις χώρες που αναφέρονται είναι χώρες που παίρνουν έτσι κι αλλιώς ε, ε, τις περισσότερες επικρίσεις ή επιφυλάξεις από το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των γεωργικών επιδοτήσεων. Ε, θα υπάρχει έλεγχος των δαπανών και της εκταμείευσης αυτών των κονδυλίων στις χώρες αυτές. Ε, στρέφομαι λοιπόν προς τη δόκτωρα Μαρίνο για την ε, απάντηση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία σε βάθος μελέτη όσον αφορά ε, τα, το ζήτημα αυτό έγιναν κάποιες προτάσεις από το Συμβούλιο, στηρίχθηκαν από τον Πρόεδρο Μπαρόζο και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι προτάσεις παρουσίαζαν ιδιαίτερα επίγοντα ε, χαρακτήρα γιατί είχαμε ε, απέναντί μας ε, χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, πολλές περικοπές στους προϋπολογισμούς τους κτλ. Όσον αφορά τώρα την ίδια τη διαχείριση, βεβαίως εμείς με κανένα τρόπο δεν σχετίζουμε την απόφαση αυτή με οποιαδήποτε ελάφρυνση, μείωση των ε, ελέγχων ενισχυμένη συνεργασία ή ενισχυμένο ποσοστό συμμετοχής ε, συγχρηματοδότησης δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι θα υπάρξει ε, και ελάφρυνση των απαιτήσεων. Πρόεδρος, νομίζω ότι κάθε περίεργος βρήκε την απάντησή του και επομένως μπορούμε, εάν βεβαίως δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρεμβάσεις, να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Δηλαδή, το επόμενο σημείο είναι ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας και θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Σε 10 λεπτά θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Διάλειμμα 10 λεπτό. Σας χαιρετίζω όλους. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.